Bien, la séance est ouverte. Mes chers collègues, donc cette séance... Αγαπητοί συνάδελφοι, 100% η σημερινή μα συνεδρίαση θα αφορά τι ψηφοφορίε, τι τελευταίε ψηφοφορίε για τον προπολισμό τη χρήση 2011. Και χθε το απόγευμα... Έκανα μια συνεδρίαση συντονιστών για να δούμε τι θα γίνει με το ψήφισμα από τη μία που θα συνοδεύσει την ψηφοφορία των τροπολογιών για τον προϋπολογισμό 2011 και να εξηγήσουμε τη σημασία την πολιτική αυτών των τροπολογιών και από την άλλη τις επιπρόσθετες τροπολογίες ούτως ώστε να υπάρξει και μια, ένας πολιτικός σύνδεσμος απέναντι στο Συμβούλιο για τους επόμενους προπολογισμούς μετά το 2011. Μετά τις εργασίες των συντονιστών και των συμφωνιών που επιτύχαμε με τους ε, συντονιστές, οι δύο εισηγητές και ο υποφαινόμενος, συμμετείχαμε σε μια νέα, σε ένα νέο γύρο της διάσκεψης των Προέδρων και με βάση τα όσα υπόθηκαν χθε το βράδυ και σήμερα το πρωί, θα σας προτείνουμε τις ε, τροπολογίες των οποίων τον κατάλογο έχετε μπροστά σας. Υπάρχουν δύο δέσμες τροπολογιών οι δημοσιονομικές, εκτός συλλογής λέγονται, μη συλλεκτικές και υπάρχουν και οι τροπολογίες που αφορούν το ψήφισμα, έτσι, σε χωριστό φάκελο. Λοιπόν, Όλοι έχετε και τους δύο φακέλους ψηφοφοριών και ελπίζω και την κάρτα την ηλεκτρονική σας. Βγάλτε τις ηλεκτρονικές κάρτες, γιατί μπορεί να χρειαστεί να μετρήσουμε. Δεν θεωρώ ότι η ομοφωνία είναι δεδομένη για όλες τις τροπολογίες. Λοιπόν, πάμε καταρχήν στις μη συλλεκτικές της. Off collection στο γαλλικό κείμενο. Υπάρχει μια σειρά τροπολογιών που αφορά την δημιουργία νέων θέσεων στον προϋπολογισμό για τις δαπάνες. Μία ανακατηγορία δαπανών. Είναι μια συμβολική πρόταση που αντιστοιχεί στις νέες αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης που τις δόθηκαν από τη Λισαβόνα. Και συνεχεία έχουμε μια άλλη σειρά από τροπολογίες για τα έσοδα. Ο Σαλβαδόρ, πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Για να κάνουμε πιο γρήγορα, Πρόεδρε, σας προτείνω όλες οι τροπολογίες που θα ψηφίσουμε από την 4.500, συγγνώμη, που αφορούν τις δαπάνες δηλαδή, να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. 4.900. Euh, ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, προφορικές τροπολογίες των σοσιαλιστών. Δυστυχώς πρέπει να τις διατρέξω. Μία-μία. Η 49.00. Ο εισηγητής. Ναι. Ποια θέση έχει. Η εισηγητη Καλύτερα. Είστε υπέρ ή κατά. Κατά. Είστε κατά. Μάλιστα. Υπέρ. Α, υπάρχει προφορική τροπολογία. Τεχνική τροπολογία. Πρέπει να διαγράψουμε το σπορ, γιατί είναι 3β και δεν έχει νόημα να την προσθέσουμε στο 4900, σύμφωνα με τα όσα λένε και οι τίτλοι. Είναι τεχνική τροπολογία. Αν υιοθετηθεί η τροπολογία, γίνεται αυτόματα. Άλλε παρατηρήσει δεν έχουμε. Ψηφίζουμε τη 49.00. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Non, tu, tu tu <laughs> Oui Bon, ok. Alors, le vote est ouvert. Ψηφίζουμε, λέει ο πρόεδρο. Και θα προσθέσουμε ότι χρειάζεται πέρας ψηφορίας. 17-14 νομίζω ότι θα πρέπει ακόμη να ψηφίσουμε δύο όχι από πλευρά ΕΛΚ και ένα ναι, επομένω πάμε 18, 16 και έγκρινε την τροπολογία, ωραία, παρακάτω. Έχουμε το 4901. Να θεωρήσουμε ότι ισχύει το ίδιο αποτέλεσμα. Ωραία. Όχι. Καλά, να ψηφίσουμε η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζουμε και θα κάνουμε τις ίδιες προσθέσεις. Έναξη ψηφοφορία. Πέρας. même μένες 17-14, το ίδιο σκορ και με τις προσθήκες πάμε στο 18, 16, πολύ ωραία, τροπολογία 49-02. Ξαναψηφίζουμε. Πέρας. 17, 13, δηλαδή πάει 18, 15 αλλά εγκρίνεται αυτή η τροπολογία, τροπολογία 49.03. Να, εδώ, εδώ έχουμε τον αθλητισμό. Ψηφίζουμε. Πέρας. Πέρας. δεκαέξι. Α, λέει ο πρόεδρος. Επομένως, και τώρα πάμε στο 18-18 που σημαίνει ότι απολύτωται η τροπολογία. Ναι, το έχω μετρήσει. Θέλετε να το ξανακάνουμε. Από τι μου λένε, έχει ψηφίσει ένας πράσινος παραπάνω. Α, δεν ψήφισε. Καλά. Επομένω έχουμε τρεις που δεν έχουν την κάρτα ψηφοφορίας, οι δύο κατά, ο ένας, δηλαδή η κυρία Ντιρό, υπέρ. Άρα πάμε στο 18-18 που σημαίνει ότι απορρίπτεται η τροπολογία. Θέλετε κάτι να πείτε? Yes, Chairman, could you just clarify which are the three people who don't have their voting cards so we all know? παρακαλώ, πόσοι έχουν και πόσοι δεν έχουν Πόσοι δεν έχουν κάρτα ψηφοφοριών. Η Σιδόνια, ο Σαλβαντόρ και, και η Ντυρό. Σιδόνια, Σαλβαδόρ και η κυρία Ντυρό. Καλά. Άρα ε, πάει η 03 και πάμε στο 4904 υπέρ. Ψηφίζουμε. Έχετε, έχετε μία προφορική. Έχετε το λόγο, κυρία. Και εμείς θέλουμε να γίνει εδώ πέρα η ίδια αλλαγή για να συμφωνούν τα πράγματα με τους τίτλους. Να μπει η αναπτυξιακή πολιτική και η πολιτική προστασία και να φύγει η EAS γιατί είναι τίτλος 5 η υπηρεσία εξωτερικής δράσης για να είναι πιο σωστά τα πράγματα σύμφωνα με τον τίτλο. Je soumets. Καλά. Επομένως ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία όπως τροποποιήθηκε προφορικά. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 14 συν 2, πάει στο 16, 16 και 1, 17, επομένως με μία ψήφο διαφορά συγκέντρωσε την πλειοψηφία τροπολογία και επομένως έχουμε τέσσερις τροπολογίες από αυτή τη δέσμη που έχουν εγκριθεί και μία που απερίφθη. Και επίση να λάβουμε υπόψη ότι όλε όσε αποφασίζονται εδώ είναι δυνατόν μια πολιτική ομάδα να λαβουμε υποψη οτι ολε οσε αποφασιζονται εδω ειναι δυνατον μια δυο ομαδα να σκατεβάσει για διοργανισμό ή στην Ολομέλεια. Εντάξει, συνεχίζουμε. Για αυτές τις τροπολόγιες και είναι αυτή που έχει σχέση με τους σπόρους, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί γιατί είναι των σοσιαλιστών. Γκόρεν ισχύει αυτό. Φάρμα. Εκτός μικροφώνου. Ε, Νομίζουμε πως το σωστό είναι να πούμε πως η εγγύηση για το μηχανισμό δημοσιονομικής σταθερότητας δεν είναι μόνο για τις πληρωμές, αλλά και για τις ε, χρεώσεις. Δεν νομίζω λοιπόν πως αλλάζει τίποτα στο νόημα. Εάν το δέχεστε, να τις ψηφίσουμε μπλοκ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Από τι μου λένε, ίσως έχετε και το 49 με την αυτομή προφορική τροπολογία. Άρα Διακόπτει ο Φάρμ. Ναι. Εννοούσα και για το 7 και για το 8 να γίνει αλλαγή για τις δύο αυτές τις τροπολογίες. Ah μάλιστα, σύμφωνοι. Άρα, προσθέτοντα υποχρεώσεις και πληρωμές. Ναι, αλλά είχε ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Άρα, όλες μαζί δεν ψηφίζουμε. 49-0 5 49.06, 49.07 και 49.08. Είναι υπέρ ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Απογειές. Ευρία πλειοψηφία και επομένως εγκρίνονται όλες μαζί. Αυτά όσον αφορά αυτή τη δέσμη εκτός συλλογή εκτό των υπολείπων. Και τώρα πάμε στην συνεργασία της οφορίας για τις τροπολογίες στον το σχέδιο ψηφίσματο του εισηγητού. Bon, donc on fera la correction. Vous avez le, tous le cahier. Έχετε λάβει ε, αυτή τη λίστα ψηφορία και έχουμε την συμβαστική του εισηγητού. Ναι, Γκόρον. Συγγνώμη που διακόπτω και πάλι, αλλά έχουμε και την τροπολογία για το φόρο των συναλλαγών που δεν την έχουμε αποσύρει. En effet. En effet. μάλιστα έτσι είναι. Οπότε πριν ξεκινήσουμε να δούμε τις τροπολογίε του ψηφίσματο. Οι σοσιαλιστέ θέλησαν οι τροπολογίε να παραμείνουν όσον αφορά του ιδίου πόρου, ούτω ώστε να θεσπιστεί αυτό ο φόρο επί των ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Τι λέει ο εισηγητής. Είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Η πλειοψηφία είναι αναμφίβολα κατά. Επομένως, απορρίπτεται από την Επιτροπή μας αυτή η τροπολογία. Όμως, όπως οποιαδήποτε τροπολογία που εδώ ε, συζητείτε, εάν θέλει ο συντάκτη τη μπορεί να την επανυποβάλει στην Ολομέλη και τώρα θα ψηφίσουμε τι τροπολογίε στο ψήφισμα. Ξεκινούμε. Συμβαστική του εισηγητή. Α, κεφαλαία. Συμβαστική. Υπέρ, κατά. Ένα κατά. Αποχέ, μία εποχή. Εγκρίνεται. Όμω δεν καλύπτονται οι δύο επόμενε τροπολογίε. Ένα της Γένσεν. Υπέρ ο συγητή, ποιοι είναι υπέρ, κατά. Ευχαριστώ. απόχέ Εγκρίνεται. Άρα οι δύο καταπίπτει. Τώρα, Τρία και τέσσερα είναι ταυτόσιμε, είναι υπέρ ο συγητή. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Παρόμοια. Οι 5 και 6 είναι ταυτόσιμες. Όμως είναι κατά ο συγκητής. υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Η επτά της Αν Γένσεν είναι κατά ο συγκητής. Ποιοι υπέρ. Κάνουμε έλεγχο ηλεκτρονικό. Ψηφίζουμε. Et, et les verts, qu'est-ce qu'ils font là-dessus Τι ψηφίζουν οι πράσινοι. Είστε υπέρ ή κατά. Καλά. Πέρα τη φορείας. 20 συν και 17 συν 2. Υπέρ και κατά. Επομένως 21-19 και τροπολογία εγκρίνεται. Βέρτμαν. που προκύψε από προφορική τροπολογία. Χάγκλαντ. Πρακτικά να πω πως ε, κάποιοι νομίζω βρήκαν τις ε, κάρτες των ψηφοφοριών μόλις τους τις έφεραν που δεν τις είχαν ε, στις πρώτες ψηφοφορίες. Οπότε δεν ξέρω εάν τώρα αυτοί, τα δύο άτομα δηλαδή είναι χωρίς κάρτες ψηφοφορίας. Μπορείτε να ξαναδείτε. Ε. Καλά. Πού βρισκόμαστε, ποιοι έχουν, ε, η κυρία ωραία. Από το ΕΛΚ. Δεν έχετε κάρτες όπως πριν. Εσύ την έχεις, ωραία. Όχι, αυτό δεν αλλάζει την ψηφορία που μόλις έγινε. Κύριε Χάγκλουν, ευχαριστώ που το θέσατε. Επομένως, μόνο ο δεν έχει την ε, κάρτα. Υπέροχο αυτό. Αυτά είναι τα προνομία του συντάκτη της έκθεσης. Αυτός θα είναι ο ρυθμιστής του τίτλου. Οπότε, θα δούμε τώρα τι έγινε με την κυρία Βέρτμαν όσον αφορά εκείνη την προφορική τροπολογία. Είναι κατά ο συγητής, είναι υπέρ της τροπολογία Βέρτμαν. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρας. 15-22. 23 κατά. Άρα απορρίπτεται. Το συμβαστικό β κεφαλαίο προφορική τροπολογία και το σε γ κεφαλαίο με την προφορική τροπολογία, αν συμφωνείτε μαζί, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Επομένω, οι δύο σημαντικέ τροπολογίε εγκρίνονται. Πάμε τώρα στο 9 του κυρίου Πόρτα, αλλά και το 10 είναι ταυτόσημα. Είναι κατά ο εισηγητή. πίνει υπέρ. Ηλεκτρονική. Ψηφίζουμε τώρα και μια που κατά. Ο εισηγητή θα, προσθέσουμε μία ψήφο υπέρ. Πέρας. μάλιστα. 20 και 19 συν 1, 20-20 απορρίπτεται. 11 και 12 είναι ταυτόσιμες. Ο συγκριτής είναι κατά. Τι είναι. Υπέρ. Κατά. là il y a une large majorité pour rejeter. Άρα η ευρύτερη πλειοψηφία είναι κατά. James Ellis. Τροπολογία Ellis κατά ο συγκριτής που είναι υπέρ. Η ομάδα του κυρίου Ellis. είναι κατά ευρία ψηφία Απορρίπτεται 14. Είναι υπέρ ο συγκητής. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Εποχές εγκρίνεται. Δέλτα. Εισηγητού. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15-16 καταπίπτουν, όμως θα πρέπει να ψηφίσουμε το 17. Τρίπελ. Είναι υπέρ, είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18, πρώτος κατοσυγητής, πίνει υπέρ, ευχαριστώ, κατά, αποχές, απορριπτωση 19, Πόρτος εισηγητής. Κατά. Το 19. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απόλυτο. 20. Χάρτονγκ. Ποιοι είναι υπέρ. Ο κύριος Χάρτον, η κυρία Ανδρέας είναι κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτονται. Η 21. Γκάρδια Θάμπαλ. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 22 του Πόρτες έχει αποσυρθεί. 23 Χάρτον είναι κατά. Συγγνώμη είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Απορρίπτεται. 24 πόρτες. Δεν έχει αποσυρθεί. Κατά τη Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 25 με χωριστή ψηφοφορία. Υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα, 25. Ψηφίζουμε. Και ψηφίζουμε μία ψήφο στις κατά, πέρα ψηφοφορίας, γιατί ψηφίσταν κατά. 23 υπέρ, 17 συν 18 κατά, άρα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ, ευχαριστώ, κατά αποχές και το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. 26. Φάρμα. Η σύγκριση υπέρ, που είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27. Γένσεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 28. Βέρτμαν, συγχυτής κατά, υπέρ, ευχαριστώ, κατά, Αποχές. Απορρίπτω. Συμβαστική ε του εισηγητού. Υπέρ. Όχι, λάθος, συγγνώμη, πριν ψηφίσουμε. Έχεις το λόγο κυρίως Πόρτας. Έχω κάνει εγώ μια πρόταση για εναλλακτικό ψήφισμα που νομίζω πρέπει να την ψηφίσουμε πρώτη. Γιατί περιορίζει το πεδίο εφαρμογή. Eh, ε, Ω προφορική τροπολογία. Nous, nous pris comme méthode... Ναι, αλλά την αρχή είπαμε πρώτα-πρώτα να ψηφίσουμε τι συμβαστικέ. για να κάνουμε πιο γρήγορα. Τι συμβαστικέ του εισηγητή. Να δούμε πώ θα πάει Εάν η συμβαστική απορρίπτεται, τότε ψηφίζουμε τις άλλε. Εκτό. αν θέλετε να κατεβάσετε μια προφορή. Ναι, ναι, ναι, αυτό θέλω να κάνω, λέει ο κύριο Πόρτο. Ε, πέστε το λοιπόν. Ορίστε, διαβάστε το. Στην παράγραφο... Θα διαβάσω αγγλικά, στην παράγραφο 9. Επαναλαμβάνει πω η διαδικασία του προπολογισμού για το 2011 έπρεπε να έχει προετοιμαστεί μαζί με μία μαζί με μία μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του πολιετούς προγράμματος. Ειδικά όσον αφορά τις, ε, τους τίτλους 1α, 3β και 4 για να αυξηθούν ε, οι προτεραιότητες και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προβλέψιμες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Ως συνέπεια αυτού, η έγκριση του υπερπολογισμού του 2011 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαρτάται από μια μεγάλη αναθεώρηση των ε, δαπανών και των ε, εσόδων που θα πρέπει να προγραμματιστεί μέχρι το 2013 τέλος ζητάει από το Συμβούλιο να λάβει πλήρως υπόψη κτλ. κτλ το ίδιο. Bien, je vous remercie, Madame le rapporteur. Εισηγήτρια, έχετε το λόγο. Προσεκτικά άκουσα και δεν συμφωνώ. Χτες υπήρξε συνένεση εν μέσω των συντονιστών. Λέει η κυρία Γεντρεύσκα εκ των εισηγητών. Πρώτα πρώτα την προφορική τροπολογία ποιοι είναι υπέρ. Κόντρ. Η Γκουε. Ποιοι είναι κατά. Οι άλλες πολιτικές ομάδες. Αποχές απορρίπτεται. Επομένως τώρα έχουμε την συμβαστική χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. L'amendement 29 το 29 όμως δεν καλύπτεται και θα το ψηφίσουμε. Όμως αυτό θα γίνει σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ο εισηγητής ή οι εισηγητές καλύτερα είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, ευχαριστώ, αποχές. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Το δεύτερο τώρα. Σε αυτή την περίπτωση είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Περισσότερο είναι υπέρ. Κατά, συγγνώμη. Άρα το δεύτερο δεν περνάει. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Καλύπτεται. Τροπολογία 31. Χάρτονγκ. Είναι κατά ζητητή. πίνει υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Α, αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική F. Η σίγματα. Η συγητή, οι συγγήτριε. Πίνει υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 32. Φάρμ εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Χάρτον, η επόμενη. Ποιοι είναι υπέρ, εισηγητής, ποιοι είναι κατά, αποχές, απορρίπτονται. 34. Έλλης. Κατά εισηγητής. υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Εδώ εδιχάστησαν οι φιλεύθεροι, όπως όλοι διαπίστωσαν, 35 πόρτες. Ψήχτες είναι κατά, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 36 πόρτες, υπέρ. Α, θα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Λοιπόν, υπάρχουν εκπλήξεις. Vote est ouvert, le vote clos. Le... ψηφοφορίες. 18-21. 21 συν 1. 37 Άλβαρο. Είναι υπέρ συγκριτής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Κρίνεται. 38 φέρν περισογητής που είναι υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Το επόμενο καταπίπτει το 39. Α, όχι, συγγνώμη, το 39 το πρώτο τμήμα καταπίπτει, αλλά θα πρέπει να ψηφίσουμε επί του δευτέρου τμήματος της τροπολογίας 39 πόρτας. Κατά εξηγητής, ποι είναι υπέρ, ποι είναι κατά. Ευχαριστώ, αποχές. Απορρίπτεται. 40 άλλο. Ε, είναι κατά ο συγκητής που είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. 41. Ε, ο είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κύριο Ρικέ. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ρικέ. Και στους συναδέλφους σας. 42. Φαν. Είναι κατά ο μην ξεχνούμε ότι πρόκειται για μια προσθήκη, προσθήκη. Είναι κατά ο συγητής, ποιοι είναι υπέρ, κατά, α, αποχές, η δεξιά, προφανώς την πλειοψηφία και απορρίπτεται, ε, την επόμενη, Άλβαρο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα έχουμε μία τροπολογία του εισηγητού προφορική. Για την καταστήση εκεί που λέει 20 εκατομμύρια στην πράγμα 18, 47 εκατομμύρια. Περ, κατά. Ευχαριστώ. Αποχές, τεχνική τροπολογία, πάντως εγκρίνεται. Έχουμε άλλες τρει συμβατέ για την ίδια παράγραφο, την 44, τρίπελ, είναι κατά ο συγητή, Ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίδεται. 45 φάρμ. Δίχως την ψηφορία, ο συγκητής είναι υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα που αναφέρει ο Γενίτερ, υπέρ, κατά, αποχές και το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται με διαφορετική όμως πλειοψηφία. Το 46, πόρτας. Συγητής κατά, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 47 πόρτας. Είναι υπέρ ο Τι είναι υπέρ, κατά. 48 Άλβαρο. Κατά ο Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. είναι Άλβαρο. Είναι κατά ο Ποιοι είναι υπέρ. Πρέπει να κάνουμε λειτουργικό έλεγχο και ψηφίζουμε το 49 του κυρίου Άλβαρο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 50 τώρα του κυρίου Έλλη κατά ο συγκριτής, Πίνει υπέρ, κατά, αποχέ. απορρίπτεται, 51. Γκόραν Φάρμ, υπέρ ο συγκριτής, Πίνει υπέρ, ευχαριστώ, Πίνει κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52, τρίπελ, είναι ο συγκριτής κατά, Πίνει υπέρ κατά αποχές Α, απορρίπτεται. «53. Γκόραν Φέρν ταυτόση με την 54. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ή ο εισηγητής. Α, τώρα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Διαφορετική πλειοψηφία έχουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. 21 ψήφι υπέρ, 18 συν κατά. Υιοθετείτε. Πρόκειται για δύο ταυτόσιμες ε, τροπολογίες. Πάμε στην 55 πόρτας. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 56. Γκέραν Φέρμα. Ο εισηγήτρια είναι κατά. Υπέρ. Παρακαλώ κατά. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Γιατί πολιτικά είναι περίπλοκη. Γίνεται περίπλοκη κατάσταση. Ξεκινάμε. Πέρας. 18 υπέρ, 19 συν 1, 20 δηλαδή κατά, απορρίπτεται. 57 της Τρούπελ σε δύο τμήματα από το should μέχρι το landscapes. Ποιος είναι υπέρ. Η συγκεκριμένη είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Ποχές. Η πλειοψηφία είναι υπέρ. Δεύτερο τμήμα. Water resources. Ποιος θέλει να βάλουμε τους υδάτινους πόρους στο landscape. Η είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ όμως. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Δεκαεφτά υπέρ, 22 συνένα 23 κατά. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. 58 Χάγκλουντ. Η ήταν υπέρ. Με προφορική τροπολογία της, των φιλελεύθερων που θέλουν η τροπολογία αυτή να πάει πιο πάνω στην παράγραφο 22. Εισηγείται υπέρ. Ποιος είναι υπέρ από σας κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 59. Firm. Φέρμ. Εισηγείται κατά. Ποιος είναι υπέρ. Ψηφίζουμε τεχνικά εδώ. Έναρξη. 20 Είκοσι υπέρ, 18 συν 1, 19 κατά. Υιοθετείτε. 60. Έλγα Τρούπελ. Η ήταν κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61. Ανδρέασεν η εισηγήτρια κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62 πόρτας. Η εισηγήτρια κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 άλβαρο. Η εισηγήτρια κατά. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 Γένσεν με μία προφορική τροπολογία. Αντικαθιστούμε το Exceptional Funding for με ειδικά μέτρα υποστήριξης της αγοράς. Η συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Όχι, λάθος έκανα, δεν υπάρχει πρώτο τμήμα. Ήταν απλή προφορική τροπολογία. Απορρίπτεται. Πάμε στην 64 Helga Truppel. Η συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ πράσινη, απομονωμένη όμως, κατά. όλα τα άλλα χρώματα κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. 66 Γκέραντ Φέρμα. Η κατά. Υπέρ παρακαλώ, υπέρ. Αϊ, αϊ, αϊ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 17 υπέρ, 22, 23, 22 σε 1, 23 κατά, απορρίπτεται. 67 Χαρτόγκ. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Je Απορρίπτεται. 68. Χατζημαρκάκης. Η ίση ήταν υπέρ. Υπέρ, παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μόνο οι σοσιαλιστές αποχές υιοθετείται. 69. Φέρμα. Ισχύει κατά. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Για την 69. Ε, Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισε και η Γιούτα. Πέρας. Αποτέλεσμα. 19 υπέρ, 20 συν 1 κατά, απορρίπτεται επομένω. 70. Χέλικα Τρούπελ. Εισηγείται κατά. Αλλά θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα την 70 ηλεκτρονικά. Έναρξη. Πέρας. Suspense. 20 υπέρ 20 και 1, 21 κατά. Απορρίπτεται. Μπράβο, μπράβο Χέλγκα. καλά τα πήγε. Ενθαρρυντικά. Θα δούμε τώρα αν η 71 θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Η συγκέντρια είναι πάλι κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία πάλι. Μια δεύτερη ευκαιρία στη Χέλγκα ας δώσουμε. Μου λένε δεν έχω πια δικαίωμα ψήφου. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 19 σημεία κατά. Αχα, περνάει. Μπράβο, Χέλγκα. Υιοθετείτε 71. Πάμε στην 72 πόρτα Η συγκέντρια είναι κατά. Υπέρ. ποιο είναι υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 73 γκερανθέρμ, η συγκέντρια είναι κατά. Υπέρ. Ελεκτρονικά το ελέγχουμε. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. 19 με 19, αλλά 19 υπέρα, 19 σαν 20 κατά, απορρίπτεται. 74, Σιμάνσκι, η ήταν υπέρ. Υπέρ παρακαλώ, ποιος είναι. Κατά. Οι σοσιαλιστές, αποχές, υιοθετείτε. 75, Helga Τρούπελ, η είναι κατά. Υπέρ, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ouvert. Sur le 75. Je ne vote pas. Ε, δεν ψηφίζω. Δεν ψηφιζω περα Πέρα ψηφοφορίας. 20-20. 20-20. Συν ένα. τέλο πάντων, όπω και να είναι, αυτό πάει να πει ότι απορρίπτεται. Τώρα πάμε στο 76 του κυρίου Άλβαρο. Ο εισηγητή είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 77 Άλβαρο. Όμω σε αυτή την περίπτωση είναι κατά ο εισηγητή, ποιοι είναι υπέρ, ηλεκτρονική ψηφορία για το 77. Πέρας. 21, 19, συν 1, 20, 21-20, άρα εγκρίνεται αυτή τη φορά 78 πόρτα, 100 ηγητής είναι υπέρ. Ε, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 79 φάρμ. Είναι υπέρ ο ηγητής, είναι υπέρ, κατά, αποχές, α, εγκρίνεται. 80 φάρμ. Είναι επίσης υπέρ ο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81. Χάρτονγκ. Κατά. Προσήγηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Πόρτος. Κατά σου ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Point de Ferme. Le rapporteur est pour. Qui est pour Merci. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 είναι συμβατή με το 83 είναι της αν γέννησεν υπερησυχτής υπέρ κατά αποχές επίσης συγκρίνεται 85 φάρμ είναι υπέρ ο συγκριτής πει είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το 86 απορρίπτεται ε, συγγνώμη έχει αποσυρθεί το 87 της Triple βρίσκεται κατά τον εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Παρά την προσπάθεια της Γκουε, δεν πέρασε αυτή η τροπολογία. τώρα στο 88 του κυρίου Κασουλίδη και του κυρίου Μπέγγεν υπέρ, ο εισηγητής ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 89 πόρτας, είναι κατά ο εισηγητής ποιοι είναι υπέρ, κατά, Αποχές. απορρίπτονται Ο 90 Βέρτμαν είναι κατά ο Σίδης, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται παρά παρά τις προσπα... την υποστήριξη της αντιπροέδρου μας, 91 γκριλίε είναι υπέρ εισηγητής, είναι υπέρ, είναι κατά αποχές, εγκρίνεται. 92 Έλλης είναι κατά. Ο συγκεκριτής ποιν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93 Βόν είναι υπέρ. Ο συγκεκριτής ποιν υπέρ. Κατά. Α, πρέπει να κάνουμε έλεγχο ηλεκτρονικό. 93 υπενθυμίζω. Υπέρ ο εισηγητής. Α, όχι, συμπάθαμε λέει ο Πρόεδρος. Διότι αλλάξαμε τη μία του προπολογισμού, άλλαξε και ο εισηγητής. Η εισηγήτρια τώρα είναι η Σιδόνια. Και βλέπω ότι είπατε κατά. Αλλάζει, αλλάζει, αλλάζει. Γυρίζουμε σελίδα. Είναι υπέρ η εισηγήτρια του 93. Όμως από ό,τι φαίνεται έχουμε περίπου ισοψηφία, άρα έχουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Δα, δα. Είναι παροτνού. 20, 20 απορρίπτονται. Je peux voter Alors maintenant je peux voter. Donc du coup, Sidonia ne vote plus. Très bien. Donc... Άρα η κυρία Γεντρεύσκα δεν είναι πλέον εισηγήτρια. Και η γνώμη της επομένως δεν ενδιαφέρει. Άρα ρωτάμε τον, τον Καρίγα μάλλον. Πάμε στο 94. Βον. Κατά συγητής. Υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Il n'y a plus de correction à faire. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα προ τα αφαιρέσει. Επομένω, από ό,τι λέει εδώ το σκορ 17-25 απορρίπτεται. 95, ε, Φαν Ντάλεν και Βοκρό. Δεν ξέρω τι πρεσβεύει ο εισηγητή, η εισηγήτρια μάλλον, free vote, κατά συνείδηση. Και... Επα... Βεβαίω, ε, επαφή με τη σοφία τη Επιτροπή. <laughs> bon, mais bien entendu, le Καλά. Ο πρόεδρός σας πρέπει να είναι ουδέτερος όμως. Ποιοι είναι υπέρ αυτή τη Τροπολογία επί της οποία είπε ότι μας αφήνει ελευθέρους η συγκέντρια. Ποιοι είναι κατά αποχές. Εν τη σοφία της η Επιτροπή μας απορρίπτει την τροπολογία. Κύριε Έλλη. Θέλω να πω κύριε Πρόεδρε, για την επόμενη ξέρω πώς θα απορριφθεί γιατί η συγγήτρια είναι κατά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να συμβιβαστούμε με το πόσο αυξάνεται το κόστος των γραφείων μας στα κράτη-μέλη, που είναι αναχρονισμός πλέον στον 21ο αιώνα και κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε. Remarque. Donc 96, le rapporteur est contre. 96 κατά. Η συγγήτρια ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97. Έλλης. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή και πάμε στο 98. Βον. Ο, η εισηγήτρια είναι κατά. Η υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99. Πώς. Τι 99 τι έχουμε. Στο 99 της Βέρτμαν έχουμε προφορική τροπολογία του κυρίου Άλβαρο. Λαμβάνουμε την ε, πρόθεση της εισηγήτριας, αλλά ίσως θα μπορούσε να συμφωνήσει να πούμε αντί για απαιτεί, ζητά. Madame Βέρτμαν fait comprendre qu'elle est d'accord de remplacer. Λέει πως συμφωνεί η κυρία Βέρτμαν να πούμε ζητά αντί για απαιτεί, είναι πιο διπλωματικό. Τι άποψη έχει ο συγγητής, είναι υπέρ. Ποιος... Πέρα αυτής της συγγήτριας με την προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Εκατό. Βόγκεν. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Ποιο είναι. Κατά. Αποχές Υπάρχει ένα μετεωρολογικό φαινόμενο πολύ ενδιαφέρον. Εξαφανίστηκε το ΕΛΚΑ. Εξαφάνιση του ΕΛΚ. Η γραμματεία μου επιβεβαιώνει ότι κάθε δεν υψώθηκε. Ίσως υπάρχει ένα σύννεφο μεταξύ των εδράνων σας και του Προεδρείου. Δεδομένου αυτού του μετρολογικού φαινομένου υιοθετείται ευτροπολογία. Θα τα ξαναδούμε στην Ολομέλεια με αυτήν την τροπολογία. 101. Ανδρέασεν. Ελεύθερη ψήφος. Επαφιέμεθα στην σοφία της Επιτροπής. Υπέρ παρακαλώ. Τώρα έχουμε αναταράξεις στους σοσιαλιστές. Άλλο μετρολογικό φαινόμενο. Πέντε δευτερόλεπτα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα παρακαλώ. διαπιστώνω το εξή. Χωρίς να θέλω να κάνω πολιτικά σχόλια, διαπιστώνω ότι όταν επικαλούμαστε τη σοφία της Επιτροπής, μπερδεύονται τρομερές σοσιαλιστές. Τα χάνουν. Ουδέτερο είναι το σχόλιο, έτσι, πολιτικά. Ποιο είναι υπέρ της τροπολογίας Ανδρέασεν. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Α, τα πράγματα ξεκαθάρισαν. Απορρίπτεται η τροπολογία. James. Αποσύρω την 102. Γιατί ο κύριος ε, Μπόκρος δεν είναι εδώ και εγώ δεν συμφωνώ. Την αποσύρω λοιπόν. Υπο, ε, απορρίπτεται την ε, υπογραφή σας. Απορρίπτεται την ίδια, αποσύρετε συγγνώμη την ίδια τροπολογία. Α, ναι, την αποσύρετε. Πολύ ωραία, τώρα το κατάλαβα. Πάμε στην 103 πόρτα. Υπέρ. Α, υπάρχουν δύο τμήματα εδώ, μισό λεπτό. Πρώτο τμήμα. Υπέρα παρακάτω πρώτα τμήματο. Κατά. Αποφέ. Απορύπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Ησίγη κατά. Υπέρ. Α, υπάρχουν δύο τμήματα εδώ, μισό λεπτό. Πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ του πρώτου τμήματο. Κατά. Αποχές. Η... Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Εισηγείται εν κατά. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται επίσης. Τέλος. Τροπολογία 83. Ε, Προφορική τροπολογία του, της εισηγήτριας, η οποία έχει μοιραστεί. Εισηγήτρια, παρακαλώ. Ναι. Θα ήθελα να διαβάσω αυτή την προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 83 υπενθυμίζει πως κατά την φάση των εκτιμήσεων και τη διαδικασία συνδιαλλαγής μεταξύ της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού και του Προεδρείου είχαμε σκεφτεί το ποσό των 1,2 ε, εκατομμυρίων ευρώ για το επίδομα γραφείου, το οποίο μειώθηκε στο 0,4 εκατομμύρια. Επενθυμίζει επίσης πως τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με το επίδομα γραφείου μπορούν να επιστραφούν μόνο κατόπιν παραστατικών, τα οποία θα δικαιολογούν το κόστος. Επισημαίνει πως οι άλλες αυξήσεις ε, που, στη σύγκριση με το έτος 2010 ε, αφορούν κυρίως ε, τα είδη εκπροσώψεις για τις υπηρεσίες ε, πρωτοκόλλου. Οπότε αν υπάρχουν αυτά τα, αν ανανεωθεί αυτό το στόκ μπορεί να υπάρξει μείωση στα επόμενα χρόνια. Επίσης τονίζει την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία όσον αφορά τις αποστολές μεταξύ των ε, εδρών εργασίας του Κοινοβουλίου και άλλων τόπων, ειδικά σε αυτούς τους καιρούς κρίσης. Οπότε καλωσορίζει την μείωση εάν τη μείωση αυτών των δαπανών σε σχέση με την πρόβλεψη που υπήρχε. Ακούσατε το κείμενο ε, από τη Χέλγα και το έχετε και μπροστά σας. Ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ. Ζητάμε χωριστή ψηφοφορία Πρώτη παράγραφος, από το recalls that μέχρι coming years. Και το υπόλοιπο είναι το υπόλοιπο του κειμένου βέβαια. Το ΕΛΚ ζητάει χωριστή ψηφοφορία για τις δύο αυτές παραγράφους, έτσι που ακούσατε. Έχετε όλη την προφορική τροπολογία για την πρώτη παράγραφο της ε, εισηγήτριάς μας, ποιος είναι υπέρ. Το... Ε, oui, alors vote électronique directement, hein, sur le... ψηφοφορία για την πρώτη παράγραφο. έναρξη, πέρας, 21 υπέρ, 17 κατά, υιοθετείται η πρώτη παράγραφος. Δεύτερη παράγραφος που προτείνει η συγκήτρια υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, υιοθετείται με άνετη πλειοψηφία. Τώρα, τώρα, έχουμε τελική ψηφοφορία για την έκθεση όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω. Έναρξη. Όλοι ψήφισαν. Πέρας τις ψηφοφορίες 36 υπέρ, 2 κατά, 4 αποχές. Θερμά συγχαρητήρια στις δύο εισηγήτριες. Έβγε. Bien, ben mes chers collègues, Πολύ ωραία. Και τώρα αγαπητοί συνάδελφοι, τα καταφέραμε στο, στο διάστημα που προεβλέπω. Α, μην πάτε που πάτε που πάτε. Δεν πάτε πουθενά χέρι όπως καταφέραμε έλεγα να καλύψουμε με αυτή την ψηφορία μια προστιθέμενη αξία σε σχέση με τα όσα είπε η διάστημα πρόεδρο. Να, ένα βήμα προς τον μπρος και άρα θα πρέπει αυτό να μας χαροποιεί και τώρα έχουμε άλλη μια ψηφορία. τον διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 3 της χρήσης του 2010 του οποίου είναι εισηγητής ο Λάσλο Σούριαν. Όλοι έχετε λάβει την λίστα για την ψηφορία. Κύριε εισηγητά θέλετε το λόγο. Yes, for I should like to... Θα ήθελα να προτείνω ψηφοφορία unblock δεδομένου του ότι ο εισηγητής υποστηρίζει όλες τις τροπολογίες. Αν συμφωνούν και οι άλλες ομάδες να το ψήσουμε μπλοκ. Όχι. Από ό,τι λένε οι φιλελεύθεροι όμως θέλουν κατά διαίρεση ψηφορία. Τι, τι θέλετε, όχι. Α, καλά. Καλά. Έλα Και τώρα. Θα ψηφίσουμε μαζί και τις οκτώ προπολογίες που αφορούν το σχέδιο διορθωτικού προβλήσμου περθών 3 πει είναι υπέρ. Κάτα. Αποχές. Οι τροπολογίες εγκρίνονται όλες μαζί. Τελική ψηφοφορία σε σχέση με το κείμενο, τον προπολισμό όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά αποχές. Δύο κατά καμία αποχή. Όλοι οι υπόλοιποι υπέρ εγκρίνονται. Και τώρα Τώρα πάμε για να ψηφίσουμε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τίτλος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε ε, τον Βόλτερ Τιερή που έχει δει στο λόγο και, ό, και όλα το Σούριαν που είναι ο συνεισηγητής έχετε το σουρίον που ειναι Σούριαν. το λογο Σουρίον. Προτείνω να ψηφίσουμε τις δύο τροπολογίες ως παράρτημα τις δύο γνωμοδοτήσεις, με συγχωρείτε, να τις ε, δεχτούμε ως παράρτημα της έκθεσης. Bien. Ε, c'est la procédure normale. Les opinions sont, Συνήθις ε, διαδικασία αυτή της γνωμοδοτήσεις τις βάζουμε, τις επισυνάπτουμε ως παράρτημα. Λάσλο. Και πάλι όμως, εάν το δεχτούν οι άλλοι, προτείνω ψηφοφορία unblock δεδομένου του ότι οι συγητές είναι κατά όλων των τροπολογιών στο διατακτικό. Γιατί είχαμε συμφωνήσει πόσο τροποποιητικός αυτός ε, προϋπολογισμός θα περάσει χωρίς ε, τροπολογία. Το κομμάτι δε, της ε, γνωμοδότησης συμφωνώ να περάσει εμπλοκ και ελπίζω να έχουμε θετική, θετικό αποτέλεσμα. Να πω και κάτι άλλο. Οι ιδέε αυτές, αυτά τα οποία πρότεινε η Ινγκε Γκρέσλε, δεν είναι κακές, αλλά ελπίζουμε στη διαδικασία της απαλλαγής ε, να μπορέσει να τα περάσει. Αλλά όχι εδώ πέρα, γιατί θα μπλοκάρει όλη τη διαδικασία. Ε, Άκουσα τους δύο εισηγητές και θέλω να ψηφίσουμε on block τις πέντε τροπολογίες για τον προπολογισμό. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Για το ψήφισμα τώρα. Θεωρούμε ότι όλες οι παράγραφοι αύκο λαμβάνονται υπόψη. Να το επαληθεύσω. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Όντω, λοιπόν, το κείμενο της Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλύπτεται. Τώρα, μένουν οι τροπολογίε κοντ, ελέγχου του προπολογισμού, το ίδιο θεωρούμε ότι λαμβάνονται και αυτές οι τροπολογίε υπόψη. Ποιο είναι υπέρ αυτή τη ιδέα, κατά, αποχέ, ναι, λαμβάνονται υπόψη. κατά, αποχέ, ναι, λαμβάνονται υπόψη. Τελική ψηφοφορία, υπέρ, υπέρ, κατά. Δύο, δύο κατά, αποχές, δεν υπάρχει εποχή όπως προηγουμένως ομοφωνία με δύο κατά και καμία αποχή. Très bien. Je Σας ευχαριστώ. Ingeborg Gressler ζητάει το λόγο για να μας παρουσιάσει το σημείο για τη διαπραγμάτευσή της για την χρηματοδότηση υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Πέντε λεφτάκια ακόμα για να ακούσετε την Ίγκε θα μας εξηγήσει λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Οι διαπραγματεύσεις, δηλαδή τι πάνε να πει διαπραγματεύσεις. Μέχρι τώρα είχαμε συναντήσει σε τεχνικό επίπεδο και ασχολούμασταν πάντα με το να εξηγούμε τροπολογίες και τους λόγους για τις τροπολογίες. Ο συνάλφος Ριβελίνη και εγώ είχαμε πολύ συγκεκριμένη εντολή. Η να ακολουθήσουμε δηλαδή τις ε, τροπολογίες ε, τις οποίες είχαμε ψηφίσει εδώ πέρα. Με ελαφρώς χαοτικό τρόπο. Και βεβαίως στόχο είχαμε να τις περάσουμε όλους, όλες και να εξηγήσουμε γιατί ψηφίστηκαν. Είπαμε πως ε, σε κάποιες δεν ήταν ξεκάθαρο το κείμενο της Κομισιόν και κάπου θέλαμε διευκρινήσεις, κάπου έγιναν αυτές. Το ίδιο το Συμβούλιο μέχρι τώρα επίσης δεν είχε τοποθετηθεί σε ορισμένες από αυτές. Ε, χτες συνεδρίασε λοιπόν η Κορεπέρ και ε, στην, Επιτροπή αυτή το αποτέλεσμα ήταν πως ε, έχει κάποιες επιφυλάξεις για 4 με πέντε τροπολογίες το Συμβούλιο, οι οποίες όμως μπορούν να αρθούν, θα έλεγα. Ε, στις δούμε με τη σειρά σε μια τροπολογία του Ρομπέρτο Καλτιέρη που είναι πάρα πολύ σημαντική αφορά την δημοσίευση των δαπανών στην εξωτερική πολιτική. Εκεί πέρα θα βρούμε μια λύση με το Συμβούλιο. Εντάξει, είναι κάπως επιθετικό το κείμενο αυτό το ομολογώ, αλλά θα βρούμε μια λύση για να λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες από ό,τι τώρα και με τρόπο κατανοητό στο παράρτημα του υπερπολογισμού ιδιαίτερα δύσκολη για νομικούς λόγους αποδεικνύεται το θέμα της ευθύνης των επικεφαλής των αντιπροσωπείων των Ευρωπαίων διπλωματών. Η κατασκευή αυτή, αν θέλετε, που σημαίνει πως οι επικεφαλής των αντιπροσωπείων προέρχονται από τις ε, εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες και εκεί θα επιστρέφουν. Οι υπηρεσία, Οπότε στο ενδιάμεσο όμως είναι ένας Ευρωπαίος ε, υπάλληλο και με ό,τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει όμως εάν, μπορούμε, εάν ανακαλύψουμε κάτι εκ των υστέρων όταν αυτός ο άνθρωπος πλέον έχει φύγει και προστατεύεται από ασυλία. Οπότε εδώ πέρα προσπαθήσαμε με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να βρούμε μια λύση η οποία θα είναι σύμφωνη και με το καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης γιατί υπάρχει μια ανάγκη καλύτερης διαφύλαξης των οικονομικών σφαιρών της κοινότητας. Γιατί σε αντίθεση με τους λοιπούς συμβασιούχους που δεν έχουν βεβαίως πολλά ποσά της Κομισιόν στη διάθεσή τους, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλα ποσά στη διάθεσή τους λόγω ακριβώς της ε, θέσης, της θέσης τους. Οπότε αντιλαμβάνομαι βεβαίως ε, τι ε, νομικέ επιφυλάξει του Συμβουλίου, αλλά χάρηκα για το ότι αναγνώρισε και το Συμβούλιο ότι έχουμε δίκαιο. Δεν καταλήξαμε τελικά όσον αφορά την ουσία. Με τον εσωτερικό ελεγκτή είπαμε πως θέλουμε από κοινού με την Κομισιόν όσον αφορά και την τήρηση των βιβλίων κάποιες επιτυχίες, σε πάση περιπτώσει, κάποια πρόοδο. Συζητούμε για το τι θα μπορούσε να γίνει. Κοιτάξτε, Υπάρχει βεβαίως αυτό το οποίο είχε πει και το ίδιο το Συμβούλιο και το οποίο ζητάει η Επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού, δηλαδή να υπάρχει αυτή η ουδετερότητα, να μην επηρεαστεί ο προϋπολογισμός, είναι κάτι το οποίο έχει αποδεχτεί ενδιάμεσα και το Συμβούλιο. Είναι δύσκολο βεβαίως, αλλά προχωράμε και βεβαίως δύσκολη κατάσταση με το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, ξέρετε, εμεί δίνουμε απαλλαγή, αλλά δεν είναι δικά μας τα λεφτά και βεβαίως ε, από εκεί που αναμέναμε τη μεγαλύτερη αντίσταση ε, όλοι, όλες αυτές οι χώρες συμφώνησαν για να συμπεριληφθεί το Κοινοβούλιο. Μιλάμε τώρα με κάποια κρατημέλη, είπαμε πως εμείς ούτως ή άλλως μπορούμε να δώσουμε αυτή την υπόθεση στον ε, Ράιμερ Μπέγκε για το πολιετές οικονομικό πλαίσιο, αλλά θα είναι η τελευταία φορά και πρέπει να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή η Κομισιόν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει αυτόν τον προπολογισμό στην πρότασή τη και να διαβεβαιώνει το, να μας διαβεβαιώσει το Συμβούλιο ότι δεν θα αναβληθεί αυτό για του Αγίου ποτέ. Πρέπει να το συζητήσουμε κάποτε και από ένα κράτο μέλο υπάρχουν σοβαρές ε, αντιστάσεις και προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα πώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρούμε μια καλή διατύπωση. για να έχουμε και έναν στόχο έτσι κάπως ε, πιο μακροπρόθεσμο. Ξέχασα κάτι. Νομίζω πως χρειάζεται ούτως ή άλλως ο τριμερής ε, διάλογος. Δεν θα έχουμε τελειώσει μέχρι Δευτέρα. Είμαστε σε πολύ τεχνικό επίπεδο ακόμα, αλλά το τεχνικό αυτό επίπεδο βεβαίως ε, έχει πάρα πολλά θετικά γιατί ξεκαθαρίζουν και πολιτικές υποθέσεις. Ερωτηματικό είναι το θέμα το που θα δίνουν ε, λογαριασμό και μιλάω κυριολεκτικά λογαριασμό για τα οικονομικά ή πρέσβεις σε εμάς. Ε, Βεβαίω δίνουν ε, λογαριασμό στην Κομισιόν, αλλά δεν μπορεί να δώσει απαλλαγή Κομισιόν. Εμεί δεν το θέλουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Οπότε υπάρχει η αρχική διατύπωση τη Κομισιόν για μία δήλωση διαβεβαίωση, την οποία αντικαταστήσαμε μέσω μια λογική διαβεβαίωση που είναι από τον διατύπωση από τον προπολογισμό, την οποία εγώ προτιμώ γιατί το statement of assurance, η δήλωση διαβεβαίωση, είναι κάτι το οποίο έχει ελεγχθεί από ελεγκτέ. Οπότε με τη λογική αυτή αξιοπιστία, διαβεβαίωση είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δεχτούμε, αλλά ε, όχι να μας στέλνουν ένα κομμάτι χαρτί και να μας ε, ξεφορτώνονται. Θα ορίσουμε το τι θα περιέχεται εκεί πέρα, αν στείλουμε κανέναν άνθρωπο σε κανένα απομονωμένο νησί ή σε καμία χώρα στην άκρη του κόσμου. Εντάξει βέβαια να λαμβάνουν υπόψη και το τι δυνατότητα υπάρχει εκεί πέρα. αλλά το θέμα της οικονομικής διαχείρισης πρέπει να το ξέρουν, να το έχουν οι άνθρωποι αυτοί που θα γίνουν πρέσβεις, να το έχουν κατά νου ότι είναι κομμάτι της δουλειάς τους και πολύ σοβαρό. Γιατί υπάρχει μια διαφορετική εντύπωση και θα πρέπει βεβαίω και η υπηρεσία να λάβει τα, τα μέτρα αυτά για να δώσει τους, στους πρέσβες τη δυνατότητα να κάνουν αυτή τη ε, δουλειά τους. Οπότε χρειαζόμαστε ακόμα κάποιες συναντήσεις με το Συμβούλιο, χρειαζόμαστε κάποιες, κάποια μέσα διαβεβαίωσης. Εγώ θεωρώ πως ε, εντάξει μπορούμε να επιτύχουμε συμφωνία αλλά γνωρίζετε πως ε, ούτως ή άλλως δεν θα υπάρξει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Η νομοθετική μας διαδικασία ούτως ή άλλως είναι πολύ εξαντλητική και θα πρέπει να είμαστε και εμείς εξαντλητικοί. Έχω και τις ε, τροπολογίες των ε, συναδέλφων και αντιλαμβάνομαι βέβαια πως κανείς δεν θέλει να υποχωρήσει. Κάτι θα δούμε. Ευχαριστώ. Ίγκε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκάθαρα μας τα είπες και όπως μας σε Ίγκε αυτό θα είναι από τα πολλά τα οποία πρόκειται να συζητηθούν την ε, Δευτέρα στον τριμερή διάλογο, οπότε και θα υπάρξει και η ευκαιρία να τα συζητήσουμε με το Συμβούλιο, να τεθεί όσο γίνεται σε πιο ψηλό πολιτικό επίπεδο το πρόβλημα, μετά από το τεχνοκρατικό πολιτικό επίπεδο και επομένως θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Επομένως, απ' θέλετε, θέλετε κάτι να πείτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω την κυρία Γκράσλε για την παρουσίασή της στο μικρόφωνο, στο μικρόφωνο σας. Να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Γκρέσλε για την παρουσίασή της και να συμφωνήσω με τα όσα μας είπε. Πλήρης υποστήριξη λοιπόν. Α, εύχομαι επίσης το Συμβούλιο να δεχτεί να περάσει στην ε, λειτουργική του φάση αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, με θετική κατάληξη στις ε, διαπραγματεύσεις, ώστε το, η υπηρεσία αυτή να λειτουργήσει επιτέλους το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ. Καλά σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες με αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύ ωραία και μέσα πριν να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας, της Επιτροπής μας, τη Γραμματεία, διότι βοήθησαν ε, τους εισηγητές και εύχομαι σε όλους καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση, γιατί την αξίζουν. Πέρα